16. 2012 τα πρακτικά της συνεδρίας 16ης Φεβρουαρίου της διάθεσή σας υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Η Επιτροπή